Good afternoon, dear colleagues. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Please be seated. We are resuming our work. Καθίστε παρακαλώ για να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Είναι 3 και 5 ήδη. Ας αρχίσουμε με την απογευματινή μας σε διάταξη και το σημείο 16, την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται να υποβάλουμε μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συντάκτηρα της γνωμοδότησης είναι η κυρία Κίνκα Γκάλ και θα υποβάλει το σχέδιο γνωμοδότησής της επί της εκθέσεως της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων με θέμα την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να έχουμε υπόψη μας καταρχήν ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει το σχέδιο εντολή για τις διαπραγματεύσεις ε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την πρόσβαση της Ευρωπαϊ... Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα υποβάλει στις, θα διοργανώσει στις 18 Μαρτίου μία ειδική δημόσια κρόαση με αυτό το θέμα. Κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή μας και είμαστε προσκεκλημένοι όλοι μαζί με την εισηγήτρια και το σκιώδη εισηγητή. Η προθεσμία για τις τροπολογίες αυτής της γνωμοδότησης λήγει στις 25 Μαρτίου. 25 Μαρτίου, παραλαμβάνω, λήγει η διορία για την υποβολή τροπολογιών επί της γνωμοδοτήσεως. Μετά τη σημερινή παρουσίαση ε, μπορούν οι βουλευτές που θέλουν το λόγο να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε τη συντάκτρια της γνωμοδότης, την κυρία Γκάλη και μετά τη συζήτηση, τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, αν υπάρχει, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Κίνγκα Γκάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι η δεύτερη φορά που εξετάζουμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων ήταν πολύ χρήσιμη και προσπάθησα να συμπεριλάβω στο σχέδιο γνωμαδότησή μου όλα τα σημεία που έδειξαν οι συνάδελφοι. Η βασική ανησυχία της δικής μας ε, Επιτροπής ε, από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ήταν ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικό μας έργο και θα πρέπει στη γνωμοδότησή μας να αναλύσουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι θα προσφέρει στους πολίτες δηλαδή αυτή η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτά τα θέματα λοιπόν προσπάθησα και εγώ να περιοριστώ. Στην προστιθέμενη αξία δηλαδή που θα έχει για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εμείς ως Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, κυρίως θέματα που αφορούν την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Δεν είναι εύκολο βέβαια να περιοριστούμε μόνο σε αυτά τα θέματα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν δύο ερωτήματα που μπορεί να κρυθούν ως τεχνικά, αλλά θα πρέπει να απαντηθούν και να καλυφθούν στην εντολή διαπραγμάτευσης και θα πρέπει ήδη αυτά τα ζητήματα να διευκρινιστούν για να ξέρουμε προς τα που πηγαίνουμε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να καθυστερήσει η διαδικασία με την διευκρίνηση αυτών των τεχνικών ζητημάτων στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, χωρίς να καθυστερούμε παραλαμβάνω την πορεία τους, θα ζητήσουμε διαλεύκανση αυτών των θεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια υποχρέωση έδρας στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. από την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Επίσης θα αρχίσει να ισχύει και το πρωτόκολλο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει δική της έδρα στο ECHR, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δηλαδή το νομικό πλαίσιο έχει θεσπιστεί. Ποιο είναι το καινοτόμο στοιχείο της νέας διαδικασίας. Καταρχήν όλα τα κράτη έχουν κυρώσει τη σύμβαση αυτή. Το καινοτόμο στοιχείο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσχωρήσει ως νομική οντότητα αυτούσια στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό δεν θα επηρεάσει την κατάσταση των κρατών μελών ως προς τη Σύμβαση. Γιατί όσα κράτη την κύρωσαν είναι μέλη συμβαλόμενα της Σύμβασης. Πάντως, για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομική οντότητα θα έχει δική της ξεχωριστή έδρα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι κάτι που συζητούσαμε εδώ και μία δεκαετία. Έχει πολύ σημαντική πολιτική επίχυση και εμπεριέχει και ένα σημαντικό μήνυμα σε ό,τι αφορά την εμβέλεια, την εμβέλεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Κάτι που επίση είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου και θα το περιλάβω στη γνωμοδότησή μου είναι ότι αυτή η προσχώρηση θα φέρει μια νέα όθηση στα ανθρώπινα δικαιώματα, μια νέα δυναμική που θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα. Πάντως την γνωμοδότηση επικεντρώθηκα στην προστιθέμενη αξία που θα έχει προσχώρηση αυτή για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω ότι θα συμβάλλει σε ένα πιο συνεκτικό σύστημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενισχύσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η σύμβαση. Όταν η προστασία που παρέχεται στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υποδιέστερη από αυτή που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, γίνεται μια αναβάθμιση προς τις προδιαγραφές της συμβάσεως. Βέβαια ο χάρτης είναι πιο φιλόδοξος και καλύπτει και άλλα δικαιώματα και αρχές ο χάρτης προβλέπει και οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, δικαιώματα προστασίας δεδομένων, ενώ η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν επεκτείνεται σε τέτοια θέματα. Οπότε δεν θα επηρεαστεί αυτή η προστασία από την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως και ένα κοινό πεδίο των δύο συμβάσεων, της Σύμβασης και του Χάρτη η προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωση ε, θα προσφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες ένα επιπλέον μηχανισμό για την ε, ενίσχυση των δικαιωμάτων. Μπορούν, για παράδειγμα, να καταθέσουν προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από μια δράση παράληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κοινοτικού θεσμικού οργάνου κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το προγραμμίσουμε γιατί εμφανίζεται συνεχώς στη συζήτηση ότι το σύστημα αυτό δεν θα τροποποιήσει το ισχύον σύστημα και τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ούτε θα επηρεάσει την απέτηση προηγούμενης ε, άσκησης όλων των ε, προβλεπόμενων ένδικων μέσων και προσφυγών. Πρώτα θα πρέπει να εξαντληθούν ε, αυτά τα ένδικα μέσα και προσφυγές. Αυτό όμως που προσθέτει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση στο σύστημα, στο γενικότερο σύστημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι προσθέτει ένα ακόμη μηχανισμό διεκδίκηση δικαιωμάτων και άσκηση προσφυγής. Και μάλιστα αυτό ενισχύει και τα διαδικαστήρια και το Ευρωπαϊκό και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα χρειαστεί συνεργασία μεταξύ των δύο δικαστηρίων για την ανάπτυξη μιας ε, συνεκτικής νομολογίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης υπάρχει το θέμα τι θα καλύπτει η εντολή και ποια θέματα θα πρέπει να πραγματευτούν οι διαπραγματεύσεις. θα είναι το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μόνο η σύμβαση και τα πρωτόκολλα. Εγώ θα πρότεινα να γίνει προσχώρηση και στα πρωτόκολλα που έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Κατόπιν υπάρχει και το θέμα της εκπροσώπησης και συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διάφορα σώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν σημαίνει ότι με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μέλο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αλλά σε όλα τα σώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης που εξετάζονται ή πειράζονται κοινοτικά θέματα, πιστεύουμε ότι και επηρεάζονται κοινοτικα θεματα πιστευουμε Ένωση θα πρέπει να είναι παρούσα. Οπότε θα πρέπει να διοριστεί ο δικαστής που θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άποψη αυτή πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει λόγο και να συμμετέχει στη διαδικασία εκλογής του δικαστού, ιδιορισμού του δικαστού. Ίσως θα πρέπει εμείς να εκλέξουμε το δικαστή και να γίνει δεκτός ο διορισμός ε, στην ε, συνέλευση ή να υιοθετηθεί μια άλλη μέθοδος για την εκλογή του δικαστού. Πάντως αυτή δεν είναι η δική μας υπόθεση, είναι περισσότερο αρμοδιότητα της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Άλλο σημαντικό θέμα είναι να καθοριστεί το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των δύο δικαστηρίων, του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου. Παρακολούθησα πολλές συζητήσεις ε, και στην έκθεση της ε, ΑΦΚΟ. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να υπάρξει ελαστικότητα για να είναι αγαστή συνεργασία και διευρυμένος ε, και τακτικός ο διάλογος. Εγώ πιστεύω ότι τα δικαστήρια θα μπορέσουν να βρουν τον καλύτερο τρόπο για διάλογο και συνεργασία και αυτό θα διευκολύνει την δημιουργία ενός συνεκτικού νομολογικού πλέγματος από τα διαδικαστήρια. Υπάρχει το θέμα του φόρτου εργασιών του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Το δικαστήριο αυτό είναι υπερφορτωμένο, έχει τεράστιο φόρτο εργασίες και πιστεύω ότι με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το σύστημα μπορεί να βελτιωθεί προκειμένου να ελαφρυνθεί λίγο το, ο φόρτος του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Ίσως θα πρέπει να πρετανεύσει εδώ και η αρχή της επικουρικότητας και τα εθνικά δικαστήρια να ε, επιληφθούν των αποφάσεων σε πρόορες φάσεις της διαδικασίας για να αποφευχθούν επανειλημμένες προσφυγές στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Πιστεύω ότι έτσι θα ανακουφιστεί κάπως το δικαστήριο του Στρασβούργου, θα απαλλαγεί από ένα τμήμα των υποθέσεων. Σημαντικό είναι να βρεθεί ισορροπία από την πρόσβαση σε ένα επιπλέον ένδικο και προσφυγή και της ανάγκης να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του δικαστηρίου. Να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο ζητουμένων. Πάντως η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση αυτή θα συνεπιφέρει και μία μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κάτι που θα ευνοήσει τους ή άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Μάλιστα, άλλου προσχώρηση στη συνθήκη δεν αφορά μόνο τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω να γίνουν διαβουλεύσεις και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συμμετέχει σε όλες τις φάσεις διαπραγμάτευσης. Επίσης να ενημερώνεται διεξοδικά για την πορεία των διαπραγματεύσεων, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες και νομίζω ότι λογικό είναι να διεκδικήσει ανάμειξη σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Σας ευχαριστώ. Αυτή ήταν μια σύντομη παρουσίαση της γνωμοδοτησής μου. Uh, Περιμένω τώρα με ανυπομονησία τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Ευχαριστούμε κυρία Γκάλ. Εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα από κάθε άποψη και από τεχνική και από πολιτική. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και δυσκολίες, αλλά σίγουρα το θέμα είναι συναρπαστικό για την πρόκληση αυτή που θα έχουμε για το επίτευγμα να αποκτήσουμε πλήρη δικαιώματα μέλους στην σύμβαση και να ισχύσουν τα δικαιώματα αυτά με τον ίδιο τρόπο σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν ανοίξουμε τη συζήτηση, να δούμε αν η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θέλει να σχολιάσουν ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Παρόλο που με είχατε συνηθίσει από την προηγούμενη, τη Σουηδική Προεδρία. Τώρα δουλεύω για την Γραμματεία του Συμβουλίου και μου ζήτησε η Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους τους. Τελευταία στιγμή είχαν κάποια άλλη υποχρέωση και δεν μπορούσαν να παρευρεθούν. Η Προεδρία επίσης μου ζήτησε να σας μεταφέρω το γεγονός ότι το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή περισσότερο βρίσκεται στη φάση της ακρόασης, της παρακολούθησης των όσων συμβαίνουν. Παρακολουθούμε τις εκθέσεις που ετοιμάζεται το Κοινοβούλιο, την διαπραγματευτική εντολή που θα υποβληθεί από την Επιτροπή και θέλουμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή διότι δεν έχουμε ένα κοινό στόχο. Ο στόχος αυτός αναφέρεται και στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Δηλαδή, πρέπει να πετύχουμε ταχεία προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό η Προεδρία είναι αποφασισμένη να το επιδιώξει και να το πετύχει όσο το δυνατόν συντομότερα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, με ιδιαίτερη χαρά να σας ανακοινώσω ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων ενέκριναν το πρωί μόλις μια σύσταση προς το Συμβούλιο με σκοπό να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Έχει μεταφερθεί εντολή αυτή ήδη στο Συμβούλιο και το σχετικό έργο στο Συμβούλιο, στο σχηματισμό του Συμβουλίου, θα ξεκινήσουν από την επόμενη Δευτέρα. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τον συνάδελφο. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την επικοδομητική μορφή της συζήτησης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε την Επιτροπή. Πολύ καλά τα νέα. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Πρώτη κυρία Κίνιγκανς. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπένοβα, ω και όντω εισηγήτρια, θα σχολίαζε κανονικά την έκθεση αυτή, όμω δεν μπόρεσε να βρίσκεται μαζί μα. Γι' αυτό μου ζήτησε να μεταφέρω την δική τη τοποθέτηση. Λέει ότι το σχέδιο έκθεση που ε, υπέβαλε η κυρία Γκάλ πολύ σωστά παρουσιάζει τι προκλήσει και τι αλλαγέ από αυτή τη νομική πράξη. Θέλει ένα πολιτικό και θεσμικό μήνυμα για την ενδυνάμωση των σχέσεων ε, της Ευρωπαϊκής, των ε, οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την υπόλοιπη Ευρώπη και βεβαίως την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την επικράτεια. Δεν θα είναι αυτή μια, η προσχώρησή μας μια απλή συμβολική πράξη, αλλά προκύπτει και μια υποχρέωση, ένας νέος μηχανισμός για να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών να μπορούν να υποβληθούν ε, και οι προσφυγές στο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο νέος αυτός μηχανισμός θα ωφελήσει ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες σε σχέση με ευρωπαϊκά νομοθετήματα. Και πολλές φορές δεν μπορούν να εξεταστούν οι προσφυγές τους από τα εθνικά δικαστήρια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η κυρία Μπένοβα ήθελε να υποστηρίξει και την κοινωνική διάσταση του θέματος αυτού, δηλαδή η κοινωνική χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι κάτι που θα λάβουμε υπόψη μας κατά την προσχώρηση στην ε, χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε τη θέση μας με αυτό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης μάλλον. Απλώς δεν βλέπει πώς άμεσα θα μπορούσε να συμμετάσχει το Ευρωκοινοβούλιο και να γίνει συμβαλόμενο μέρος στην ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση καθότι το, η προσχώρηση αυτή δεν ε, σημαίνει την αυτόματη προσχώρηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν δύο ξεχωριστοί οργανισμοί. Επίσης, κατά την άποψή της, θα είναι κάπως δύσκολο να έχουμε περισσότερη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα, στους φορείς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και πιθανόν να υπάρξουν και αρκετές ε, διαπραγματεύσεις και ε, ανάγκη ανταλλαγμάτων με τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν κάπως επιφυλακτική κυρία Μπένοβα και θέλει να γίνουν κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση ε, πιστεύει βεβαίω ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει δράση στην όλη διαδικασία, καθότι το θέμα αφορά τα δικαιώματα των πολιτών τη Ευρώπη και τη στιγμή που διορίζεται ένα δικαστή για το δικαστήριο στο Στρασβούργο, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επηρεάζει κατά την διορισμό και την διεξαγωγή των διαφόρων υποθέσεων. Ο κ. Λούτσεφ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνο με την εκτίμηση των προηγουμένων ομιλητών επί του σχεδίου γνωμοδότησης, τη συναδέλφου κυρίας Γκάλ. Σήμερα δόθηκε ένα καλό μήνυμα και οι συνάδελφοι στην ε, Επιτροπή ΑΦΚΟ θα ενθαρρυνθούν για να αρχίσουν όλες τις ε, προετοιμασίες για την οριστικοποίηση ε, και ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας που αναμένεται μετά από 15 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί η Ισπανική, η Ουγγρική, η Βελγική Προεδρία ε, θα είναι οι ε, Προεδρίες που θα φροντίσουν για την ολοκλήρωση του θέματος. Ε, πρέπει να επεξεργαστούμε επιπροσθέτως και άλλα κέρια ζητήματα που φωτίζονται από το σχέδιο γνωμοδότησης για να εμπλουτίσουμε τη δική μας οπτική και να βοηθήσουμε και τον εισηγητή κύριο Ατόντο, ο οποίος είναι ο εισηγητής από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Πιστεύω ότι η παράγραφη, το κείμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια διευρυμένη ε, αξιολόγηση είναι η παράγραφη 5, 6 και 8 από το σχέδιο γνωμοδότησης και ιδιαίτερα η παράγραφος 5 γιατί προσπαθεί να διασκεδάσει κάποιες ανησυχίες που έχουν σχέση με τη σχέση μεταξύ εθνικών δικαστηρίων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο και το ε, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι θα πρέπει να εμβαθύνομαι σε αυτό το θέμα. Τώρα για την παράγραφο 6. Αναρωτιέμαι γιατί αναφέρεται στην αναμενόμενη συνεργασία μεταξύ εθνικών δικαστηρίων και των δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε είτε εδώ ή στην άλλη έκθεση ε, κάτι προς την κατεύθυνση της άμεσης της ενθάρρυνσης από, τα, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ώστε να ανταποκριθούν στη βούλησή μας. Ε, καταδεικνύοντας και τη δική τους βούληση και προθυμία να επιταχύνουν την διαδικασία προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Είμαστε στις πρώιμες φάσεις της διαδικασίας, αλλά νομίζω ότι τα κράτη-μέλη έδωσαν, έστειλαν ένα μήνυμα ε, και θα πρέπει να ε, λάβουν και άλλα μηνύματα από μας σχετικά με τη βούλησή μας να φροντίσουμε για την επιτυχή προσχώρηση της Ένωσης ε, στην ΕΣΔΑ. Η παράγραφος 8 επίσης λέει ότι τεχνικής φύσεως ανεπίλητα θέματα μπορεί να δημιουργήσουν εμπόδια, φραγμούς στην ομαλή διαδικασία προσχώρησης της Ένωσης στη Σύμβαση είναι δυνατόν να παραθέσουμε κάποια από αυτά τα τεχνικά θέματα, γιατί ίσως κάποια έχουν σχέση με την εκπροσώπηση της Ένωσης ε, στα σώματα του Συμβουλίου. Ίσως να είναι διαφορετικής φύσεως. Καλό θα ήταν να αναφέρομαι κάποια τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε στη διαδικασία της προετοιμασίας για την προσχώρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Ρωμέβα. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα, ελάχιστα έχω να προσθέσω, γιατί τα πιο σημαντικά ετέθησαν ήδη και πρέπει να ζητήσω και συγνώμη γιατί ο πραγματικός σκιώδης των Πρασίνινων, ε, κυρία Χάουταλα, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Ένα θέμα θέλω να θέσω που νομίζω ότι είναι κέρια σημασίας ε, και πρέπει να το διευκρινίσουμε ως θέση του Κοινοβουλίου. Αφορά το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο της εφαρμογής. Νομίζω ότι δεν συζητήσαμε ότι πρέπει να αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το επίπεδο εφαρμογής. Νομίζω ότι δεν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να εφαρμόζεται και να ισχύει και για όλες τις εξωτερικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν είναι τουλάχιστον στο Συμβούλιο τόσο σαφές αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Διαβάζοντας την έκθεση δεν το βλέπω είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δεν αναφερόμαστε μόνο στα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης, αλλά λαμβάνουμε υπόψη και όλες τις δραστηριότητες παγκοσμίω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ομολογώ ότι δεν ξέρω πώς θα ε, ενσωματωθεί αυτό στο κείμενο, δεν το έχω βρει, ίσως ε, η συγγήτρια μπορεί να μας διαφωτίσει. Ευχαριστώ. Κυρία Βέρχαρτ. Α, συγγνώμη, το, έκανα λάθος το όνομά σας. Εζιάτ. Πολλά ήδη έχουν ακουστεί. Εγώ ήθελα απλώ να επιμείνω σε κάποια στοιχεία, γιατί μου φαίνεται σημαντικά και δεν συμφωνώ απολύτω με την εισηγητριά μας, κάτι που δεν συνηθίζει να συμβαίνει, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερω το θέμα τη περιμέτρου που θέλουμε να καλύψουμε η σύμβαση, τα πρωτόκολλα της και η Ευρωπαϊκή Χάρτα. Νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το περιεχόμενο της έκθεσης ως προς αυτή τη διάσταση. Συμφωνώ με όσα είπατε, ιδίω για το θέμα των πρωτοκόλλων, όταν συνυπογράφονται από το σύνολο των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως θα μπορούσαμε ως Ευρωκοινοβούλιο να έχουμε ένα ρόλο περισσότερο ενθαρρυντικό να πούμε δηλαδή ότι θα επιθυμούσαμε το σύνολο των κρατομελών να υπογράψουν το σύνολο των πρωτοκόλων υπό την αίρεση βέβαια της ε, περαιτέρω επιφύλαξής μας και οι κοινωνικοί εταίροι για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ε, άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση είναι πολύ πιο ευρεία από ότι κοινωνική χάρτα, η χάρτα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να ξαναδούμε νομίζω το περιεχόμενο ε, έτσι ώστε να δώσουμε ένα σύνθημα, ένα, ένα, συγγνώμη, ένα μήνυμα θετικό ως προς όλες τις ε, επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν ε, από την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπουζούτηλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κίνκα Γκάλ για την έκθεσή της και για την εργασία της. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη αφορά τους πολίτες και την ανάγκη να ε, ε καλυφθούν Χαίρομαι που η κυρία Γκάλ συμπεριέλαβε ε, το θέμα αυτό, τη σημασία δηλαδή της ε, ενημέρωσης των πολιτών εξηγώντας την προστιθέμενη αξία της προσχώρησης προς όφελός τους. Επιμένω σε αυτό γιατί αν δεν πείσω με τους πολίτες ε, ότι έχουν να ωφεληθούν από αυτή τη διαδικασία, τότε θα εργαζόμεθα επιματέω, γιατί αυτό το νέο μέσο δεν θα χρησιμοποιηθεί. Και υπάρχει και μεγάλη σύγχυση, όπως και ε, παρανοήσεις. Πιστεύουν, πιστεύουν πολλοί ότι θα αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα, πράγμα που δεν θα είναι αναγκαστικά το αποτέλεσμα αυτής της προσχώρησης στη σύμβαση. Ε, δεν ξέρω εάν υπάρχει ε, κάποια προεργασία σε αυτό, ε, κατευθυντηρίες γραμμές, προγράμματα ενημέρωσης προβλέπονται, γιατί θα πρέπει να πιστούμε. Είναι σαφές ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί. Γιατί λοιπόν να μην εντάξουμε και τους πολίτες στη διαδικασία αυτή ώστε να είναι ενήμεροι. Ελπίζω η Κομισιόν να μας εξηγήσει τι κάνει ή τι προτίθεται να κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερο και τελευταίο, ε, έχω μια σύγχυση ακόμη σε σχέση με τις μελλοντικέ σχέσεις μεταξύ των δύο δικαστηρίων, το 10 και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί φοβάμαι ότι και εδώ ε, ίσως υπάρχει κάποια ε, δυνητική σύγκρουση ή σύγχυση όπου και οι δύο πλευρές θα θεωρούν ότι ε, θα έχουν τον τελευταίο λόγο η καθεμία για λογαριασμό της. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί επίσης. Επίσης, ε, για πρώτη φορά από ό,τι φαίνεται, θα υπάρχουν δικαστές που θα είναι, δεν θα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ε, συζητούν για δικαιώματα πολιτών στην Ένωση. Θα πρέπει ο εισηγητής να παρακολουθήσει πολύ το θέμα των σχέσεων μεταξύ ΔΕΚ και ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ερχόμενο σε άμεση επαφή και συζήτηση και με τους δύο, γιατί αυτή η σχέση πρέπει να διευκρινιστεί όχι για τα δύο δικαστήρια μόνο, αλλά και για μας. Η κυρία Σόφινφελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά ελέγχθησαν ήδη, δεν θα προσθέσω πολλά. Πρώτον γιατί δεν είμαι η επίσημη σκιώδης, η επίσημη ζητή συγγνώμη ήταν νωρίτερα εδώ αλλά έπρεπε να φύγει ξαφνικά. Μία παρατήρηση. Αναφέρεται στην παράγραφο 7, τέταρτη παύλα, κάνετε αναφορά στην εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και λέτε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, υποθέσεις που αφορούν και εντάσσονται στο εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να εξετάζονται από το δικαστήριο. Φαντάζομαι ε, ότι αναφέρεστε εδώ σε ε, υπερβολικό αριθμό εκκρεμών υποθέσεων κλπ. Σε πολλές χώρες πίσω από την αρχή της επικουρικότητας κρύβεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή μια αναγνώριση της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου. Πολλοί δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις του δικαστηρίου και είναι αυτές χώρες που ανοιχτά αμφισβητούν την δικαιοδοσία του δικαστηρίου σε κάποια θέματα. Θα ήταν πολύ λυπηρό αν έτσι ερμηνευόταν η συγκεκριμένη διατύπωση. Θα κοιτάξουμε μέσα από τροπολογίες να διασφαλίσουμε το σωστό νόημα και να αποφύγουμε ε, παρεξηγήσεις. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Κίνγκα Γκάλ, θα ήθελα να κάνω μια εξαίρεση στο κανόνα που έχω επιβάλει στον εαυτό μας πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, στο να παρεμβαίνω επί της ουσίας κατά τη συζήτηση, γιατί πιστεύω ότι ο ρόλος του Προέδρου είναι περισσότερο συντονιστικός ε, κατά τις συζητήσεις ε, και όχι τόσο παρεμβατικός. στη συζήτηση. Εν προκειμένου όμως υπάρχει ένα θέμα που θέλω να παρουσιάσω στα μέλη της Επιτροπής. Το θέμα αυτό αφορά το διάλογο που πρόκειται να ανοίξουμε μεταξύ ε, των δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Πάντοτε ήμουν της γνώμης ότι η προσέγγιση ε, με την οποία η συνθήκη της Λισαβόνας παρουσιάστηκε στους Ευρωπαίους πολίτες είναι μια προσέγγιση ε, που τονίζει την απλούστευση. Αυτό μπορεί να είναι και υπονομευτικό. Καλό είναι να ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλει να γίνει διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη ταυτόχρονα. Όμως πρέπει και εμείς να μαθαίνουμε για να ενημερώνουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Και ε, εδώ δεν πρόκειται μόνο για απλούστευση, αλλά και για βελτίωση. Καμιά φορά η βελτίωση δεν προέρχεται από την απλούστευση. Καμιά φορά ε, στηρίζεται στη συνθετότητα. Ε, γιατί υπάρχει και η διάσταση της συνθετότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και είμαστε ταυτόχρονα και πολίτες κρατών εθνών. Και αυτή η διπλή ιδιότητά μας δεν απλουστεύει τα πράγματα, όμως τα βελτιώνει, θεωρώ, για όλους μας. Και αυτή νομίζω σε τελευταία ανάλυση είναι η προσέγγιση που πρέπει να υιοθετήσουμε ώστε να ε, παρακολουθήσουμε τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ δικαστηρίων. Ένα δικαιικό σύστημα στηρίζεται σε μόνιμο ανοιχτό διάλογο μεταξύ δικαστηρίων. Κάθε δικαστήριο έχει ένα λόγο που μπορεί να είναι ο τελεσίδικος ή όχι εξαρτάται από τις προσφυγές, ενστάσεις, ε, οι εφέσεις ή τα ε, ε, μέσα που παρέχονται εάν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος από την απόφαση ενός δικαστηρίου. Η ερμηνεία σχετικά με την τελεσιδικία ενός δικαστηρίου ανταποκρίνεται στην ε, νομική πυραμίδα ε, ενός συστήματος εδώ, εν προκειμένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε μία πυραμίδα με ένα ανώτατο δικαστήριο που είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο αδιαμφισβήτητα, τα συνταγματικά δικαστήρια δεν δέχονται ότι το Ευρωπαϊκό ε, Δικαστήριο είναι ανώτερο δικαστήριο σε μια πυραμίδα ε, δικαιού συστήματος. Υπάρχει διάλογος με το 10 και αυτό ήδη θα ισχύσει και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ανοιχτό συνεχής διάλογος των δύο δικαστηρίων. Το 10 έχει τον τελευταίο λόγο στην ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαίου και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει τον τελευταίο λόγο στην ερμηνεία της συμβατότητας ημί κανόνων, υπράξεων που έχουν εγκριθεί ή εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα πρέπει να δεσμεύεται από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου περί της ερμηνείας της εφαρμογής της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δεν είναι ε, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ε, το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οπότε, ναι, εδώ έχουμε ε, μια, ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο δεν θα μας επιδεινώσει ε, την κατάστασή μας, ούτε θα μειώσει τα, ανθρώπινα, τα δικαιώματά μας. Αντίθετα θα τα πολλαπλασιάσει και θα τα βελτιώσει, γιατί δρά πολλαπλασιαστικά στις δυνατότητες που έχουμε για προσφυγή σε ένδικα μέσα και προστασία και ικανοποιητική νομική απόκριση ε, όταν κάποιος είναι πεπισμένος, βασίμος ότι κάποιο δικαίωμά του το οποίο διασφαλίζεται από την ΕΣΔΑ έχει παραβιαστεί από κάποιο κράτος μέλος το οποίο προσυπογράφει την ΕΣΔΑ συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν προκύψει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα ζήτημα που ήθελα να θέσω ε, στην Επιτροπή για να ε, προαγάγουμε την γόνιμη συζήτηση που θα αρχίσει και θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Καθώς θα προχωρούμε ε, στη διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξανα... Ε, δίνουμε το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Γκάλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το ζήτημα, αλλά τώρα έχουμε μπει στο χώρο. Και το σημαντικότερο είναι να καταλάβουν όσο τα δυνατόν περισσότεροι πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πάζλ. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό που είπατε και αυτό που είπε ο κ. Μπουζούτιλ ότι η Επιτροπή θα πρέπει να σκεφτεί την περίπτωση να ετοιμάσει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και μετά κατευθυντήριε γραμμέ. για το ποια θα είναι προστιθέμενη αξία αυτή τη προσχώρηση. Να μπορούν και οι πολίτε να καταλάβουν ποια θα είναι τα ωφέλη του, γιατί παραμένουν διάφορα ζητήματα εκκρεμή. Κανεί δεν γνωρίζει τι απαντήσει από τώρα. Μόλι ξεκινούμε στη φάση και περνάμε στη φάση των διαπραγματεύσεων. Όμω, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και τις ιδέες τους. Απλώς νομίζω τα περισσότερα λίγο πολύ καλύπτονται από την έκθεση. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτική για το όλο θέμα. Δεν μπορώ λοιπόν να δείξω σκεπτικισμό. Και τώρα εφόσον υπάρχει υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει σε αυτή τη σύμβαση. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να κρίνουμε το θέμα διαφορετικά. Απλώς να εξηγήσουμε σίγουρα σε όλους ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα για τους πολίτες. Και προσπάθησα να τα συμπεριλάβω όλα αυτά ήδη στα πρώτα άρθρα, στις πρώτες παραγράφους δηλαδή, της έκθεσής μου, 3, 4, 5 και 6. Τι πιστεύω εγώ ότι θα είναι τα ωφέλη για τους πολίτες. Ρωτήθηκε γιατί τα τεχνικά προβλήματα δεν απαριθμώνται. Νομίζω ότι αναφέρθηκα σε αυτά στην παράγραφο 8. Όμως περισσότερο αναφέρομαι στα εκκρεμή νομικά, τεχνικά και θεσμικά ζητήματα που αναφέρονται και αναλύονται περισσότερο στο, στην παράγραφο 7. Θα πρέπει λοιπόν να επιληθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ιδάλω δεν θα είμαστε πραγματικά σε θέση να ωφεληθούμε αμέσω από τη νέα δυνατότητα τη προσχώρηση. Βεβαίω, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, για τα θεσμικά ζητήματα δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε οι τεχνικές δυσκολίες να καθυστερήσουν την όλη διαδικασία, χωρίς λόγο. Η κυρία Χάουταλα έθεσε το ερώτημα του πεδίου της εμβέλειας. Εδώ σε αυτή την ε, έκθεση δεν ήθελα να καλύψω τους πολίτες τρίτων χωρών, διότι υπάρχει άλλη γνωμοδότηση που ετοιμάζεται, την γνωμοδότηση του κυρίου Πρέντα από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που καλύπτει ακριβώς αυτό το σημείο. Η δική μου υποχρέωση εδώ ήταν να καλύψω το ζήτημα της προσχώρησης, αλλά από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι από τη σκοπιά των τρίτων χωρών. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να δείτε τις δύο ε, γνωμοδοτήσεις από κοινού στο τέλος, ως αλληλοσυμπληρούμενες. Και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει μέχρι την ετοιμασία της τελικής έκθεσης και ότι ο εισηγητής από την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων θα συμφωνήσει με αυτή την ε, αντίληψη. Ότι ακολουθούμε δύο διαφορετικούς δρόμους αλλά για να καταλήξουμε σε κοινό προορισμό. Επίσης ρωτήσατε και αναφέρετε κάποια στοιχεία που υπάρχουν νομίζω στην παράγραφο 7 στο πρώτο εδάφιο. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπουσούτιλ όπως προείπα. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θέλω να ακούσω και τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγώ. Τι σκοπεύει δηλαδή να κάνει η Επιτροπή για να δείξει στους πολίτες τι θα κερδίσουν από όλα αυτά και για την αρχή της επικουρικότητας. Ακριβώς για να αποφύγουμε την διπλή εκδίκαση υποθέσεων το συμπεριλάβαμε αυτό. Η διάσκεψη του Interlaken αναφέρεται ακριβώς στο έργο και τις δυσκολίες του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επαναλήφθηκε πολλές φορές ότι το όλο πρόβλημα πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Εξού και στην τελική δήλωση της διάσκεψης αυτής περιελήφθηκε αυτή η παρατήρηση. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο το χρησιμοποιώ και εγώ εδώ. Για να αποφύγουμε την, την ε, πολλαπλή εκδίκαση των ίδιων υποθέσεων. Και όχι για καμιά άλλη σκοπιμότητα. Εάν τώρα έχετε κάποια τροπολογία για την καταλληλότερη διατύπωση, ευχαρίστω εάν νομίζετε ότι είναι παραπλανητική. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Περιμένω τις τροπολογίες σας. before... Ευχαριστούμε κυρία Γκάλ. Πριν θέσουμε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, νομίζω ο κύριος Κλέης θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ. Έχω μια σύντομη ερώτηση. είχα υποβάλει μία πρόταση να προσκαλέσουμε κάποιον από το δικαστήριο για να μας διαφωτίσει. Γιατί και ο κύριος Μπουσουτήλ και εγώ έχουμε απορίες και αναπάντητα ερωτήματα μετά την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του καθηγητού Ζακέλ. Δεν ε, έχουν απαντηθεί όμως όλα αυτά τα ερωτήματα, γι' αυτό και μας ενδιαφέρει η άποψη του δικαστηρίου. Οι συντονιστές ε, δεν εξέτασαν καθόλου αυτή την πρόταση. Θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, κύριε Κλέης, χθες, στη συνεδρίαση των συντονιστών, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε επίσκεψη και στα δύο δικαστήρια, και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Και φυσικά η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλα τα μέλη. Ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίε μόνο. Γιατί είναι αδύνατο να επισκεφθούμε και τα δύο δικαστήρια την ίδια μέρα, μια και το ένα βρίσκεται στο Λουξεμβούργο και το άλλο στο Στρασβούργο. Αλλά θα μπορούσαμε να το προγραμματίσουμε για 5 με 7 Μαΐου. Να κανονίσουμε δηλαδή 5 με 7 Μαΐου την επίσκεψη στα δύο δικαστήρια. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση, πάντως λήφθη υπόψη πολύ σοβαρά η πρότασή σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ευχαριστώ. Ακούσαμε με ιδιαίτερη προσοχή τα σχόλια και τα σημειώσαμε και φυσικά θα λάβουμε υπόψη τη σύστασή σας να προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώσει τους πολίτες για αυτό το σημαντικό θέμα. Βέβαια βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο αυτής της διαδικασίας προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα πρέπει να προβλέψουμε τα κατάλληλα μέτρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορέσουν να ασκήσουν τα νέα δικαιώματα και να αξιοποιήσουν τις νέε δυνατότητες που τους προσφέρει η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνθήκη, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια? Όχι. Οπότε αν όλοι συμφωνείτε, ορίζουμε τη διορία για την κατάθεση των τροπολογιών στις 25 Μαρτίου το μεσημέρι. 25 Μαρτίου 12 το μεσημέρι, λίγη η διορία για την κατάθεση των τροπολογιών. Κατόπιν θα ψηφίσουμε στην Ελευθεριών στις 27 και 28 Απριλίου. Ενώ στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε τον Ιούνιο. Συμφωνούμε με το χρονοδιάγραμμα. Πολύ ωραία και σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 17. Το σημείο 17 προβλέπει τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικέ υποθέσεις. Θα ακούσουμε την παρουσίαση από την Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου. Ξέρετε ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας προβλέπει τέτοια αμοιβαία συνδρομή. Παρακαλώ όσοι φεύγουν από την αίθουσα να μην ε, δημιουργούν φασαρία. It's been Ήταν αρκετά εκτενής η συνεδρίαση και αυτό είναι το τελευταίο σημείο της απογευματινής ημερήσιας διάταξης. Λίγη υπομονή λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. Το θέμα αυτό έτυχε διαπραγμάτευση το 2009 και η συμφωνία αυτή έχει πλέον δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόταση του Συμβουλίου που θα πρέπει να εγκριθεί. Με βάση το άρθρο 218 της Συνθήκης της Λισαβόνας χρειάζεται η συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Γιακολίνο, αλλά πρώτα στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας παρουσιάσουν το περιεχόμενο της συμφωνίας με την Ιαπωνία. Τελικά μου είπαν ότι δεν θα μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μόνο εκπρόσωπος ε, της Ισπανικής Προεδρίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε στην Ισπανική Προεδρία να σας παρουσιάσει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας με θέμα την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικέ υποθέσεις. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι στη συνεδρίασή σας για να σας παρουσιάσω τη συμφωνία αυτή. Θα ήθελα καταρχήν να σας εξηγήσω για ποιους λόγους υπεγράφει αυτή η συμφωνία. Οι λόγοι για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ήταν τρεις. Μία τέτοια συμφωνία δικαστικής συνδρομής επιφέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία στις δικαστικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλωμένων μερών. Γιατί άλλο να υποβάλλονται αιτήματα δικαστικής συνδρομής μέσω μιας συμφωνίας και μιας προκαθορισμένης οδού από ότι αν δεν υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο. Επίσης δεν υπήρχε καμία συμφωνία κανενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ιαπωνία για αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. Οπότε είτε θα αφήναμε στα κράτη-μέλη να συνάψουν διμερώς τέτοια συμφωνία ή να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία. Οπότε θα είχαμε διμερείς συμφωνίες ορισμένων μόνο χωρών μελών με την Ιαπωνία, αλλά θα υπήρχαν διαφορές ακόμη και στις επιμέρους συμφωνίες αυτές. Γι' αυτό ήταν καλύτερο να επιδιώξουμε ένα ενιαίο πλαίσιο με συμβαλόμενο μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε και η Ιαπωνία είχε ενδιαφέρον να συνάψει τη συμφωνία με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από μία δεκαετία περίπου, το, η Ιαπωνία δεν είχε συνάψει καμία συμφωνία δικαστικής συνδρομής για ποινικέ υποθέσεις με καμία χώρα του κόσμου. Βέβαια, την τελευταία δεκαετία η Ιαπωνία έχει αλλάξει την πολιτική της και έχει συνάψει τις συμφωνίες με την Νότιο Κορέα, την Ρωσία, την Κίνα, τους γειτονές δηλαδή, αλλά και με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Οπότε ξεκίνησε μια πολιτική δικαστική συνεργασίας ε, της Ιαπωνίας με τις άλλες χώρες, οπότε υπό αυτό το πρίσμα της νέας πολιτικής ε, ήταν ε, αναμενόμενο να εκδηλωθεί ενδιαφέρον και είχε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ιαπωνίας. Η συμφωνία αυτή δικαστική συνεργασία επικεντρώνεται στα πιο συνηθισμένα θέματα ποινικών υποθέσεων, παρουσίαση μαρτυριών, υποβολή αποδείξεων κτλ. Επίσης προβλέπει τη χρήση της τηλεδιάσκεψης, αλλά και η δυνατότητα λήψης ε, πληροφοριών από τις τράπεζες. Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες από τις τράπεζες, δεν ήμασταν πολύ φιλόδοξοι εξαιτία του Ιαπωνικού τραπεζικού συστήματος που δεν έχει μια κεντρική βάση που να επιτρέπει τη λήψη μιας πληροφορίας για το κατά πόσο κάποιος έχει ανοίξει λογαριασμό στην Ιαπωνία. Οπότε οι μόνες πληροφορίες που μπορούν να δώσουν οι Ιαπωνικές αρχές για τα θέματα αυτά είναι για μια συγκεκριμένη τράπεζα, για συγκεκριμένες τράπεζες να δίνονται πληροφορίες. Αλλά κεντρικό αρχείο δεν υπάρχει. Οπότε οι πληροφορίε που μπορεί να δώσει η Ιαπωνία από την άποψη αυτή είναι πολύ περιορισμένε. Στην Ιαπωνία άλλωστε υπάρχουν πάρα πολλέ τράπεζε και επειδή δεν υπάρχει κεντρική βάση, είναι αδύνατο να υποβληθεί αίτημα δικαστική συνεργασία με την Ιαπωνία ε, ζητώντα πληροφορίε ε, για συγκεκριμένου λογαριασμού ή κινήσει ενό ενός λογαριασμού, γιατί θα πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων η συγκεκριμένη τράπεζα ή τράπεζε με τις οποίες ε, υπάρχουν συναλλαγές, στις οποίες βρίσκονται αυτοί οι λογαριασμοί. Ως προς το περιεχόμενο υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που λαμβάνονται, γιατί οι πληροφορίες αυτές περιορίζονται στους, στόχου, στους στόχους για τους οποίους ζητήθηκε η πληροφορία. Δεν μπορεί η πληροφορία αυτή να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Επίσης, μας ενδιαφέρουν οι διατάξεις για τη θανατική ποινή. Όπως ξέρετε, η Ιαπωνία είναι μία από τις χώρες που δυστυχώς εξακολουθεί να ε, προεβλέπει στο σύστημά της τη θανατική ποινή. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται συχνή χρήση της θανατικής καταδίκης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται, επιβάλλεται η θανατική ποινή. Ε, αυτό ήταν ένα σημαντικό κόλλημα στις διαπραγματεύσεις που υπερκεράστηκε με ένα πολύ καινοτόμο τρόπο. Γιατί προβλέπεται ότι η δικαστική αρχή μπορεί να απορρίψει τα αιτήματα δικαστικής συνεργασίας που προέρχονται από την Ιαπωνία αν δεν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία των Ιαπωνικών αρχών που θα λαμβάνουν τη δέσμευση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθεί η πληροφορία που ζητά και που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για οποιαδήποτε διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή θανατικής καταδίκης. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι η συμφωνία είναι καλή και ως προς το περιεχόμενο και ως προς την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου. Γι' αυτό και το Συμβούλιο ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας να δώσει την έγκριση για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε απορίες σας. Ωραία. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Γιακολίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Παρακολούθησα με προσοχή τι πληροφορίε που μα έδωσε η Προεδρία του Συμβουλίου. Ευχαριστώ την ομάδα μου που μου ανέθεσε αυτή την ε, έκθεση και μου έδειξε εμπιστοσύνη έτσι. Και θεωρώ ότι μια συμφωνία συνδρομής όπως αυτή που ανέπτυξε η Προεδρία και για έναν κολοσσό όπως η Ιαπωνία με εταιρείε που είναι όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένες με σχέσεις όλο και περισσότερο εντατικές και συχνές με τα κράτη-μέλη. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Οι σχετικές δραστηριότητες ξεκίνησαν από το Φεβρουάριο του 2009. Λήφθηκε απόφαση από το Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου του 2009 και όλα είχαν αναβληθεί μέχρι την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Στο παρελθόν, οι σχέσεις συνεργασίας και η συνδρομή μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών και της Ιαπωνίας προβλέπονταν και καλύπτονταν από σχέσεις συνεργασίας όχι και τόσο συχνέ Μέσω μιας μελέτης μάλιστα που έχουμε να καλύπτει το διάστημα από το 98 στο 2007. Μόνο 556 περιπτώσεις είχαμε σε αυτό το διάστημα στις υποθέσεις με την Ιαπωνία. Να λοιπόν μια ευκαιρία να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία, τη δικαστική, την συνδρομή, που ούτως ή άλλως ρητός προβλέπει και η συνθήκη της Λισαβόνας και την επικυρώνει. Επίση προβλέπονται και συγκεκριμένε δυνατότητες όπου υπάρχει απέτηση αναστολής της ε, συνεργασίας η παραπομπής σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, ανάλογα με τις έρευνες που γίνονται, η διαδικασία παραπομπής περιγράφεται με λεπτομέρειες, φαίνεται αρκετά απλοποιημένη, ήδη αναπτύχθηκαν τα αίτια άρνησης ή απόρριψης, Υπάρχουν και κάποιες νέες ευκαιρίε σε σχέση με την τηλεδιάσκεψη. Επίσης αναφέρατε και το άρθρο 18 για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και το αναπτύξατε. Οπότε νομίζω ότι η εμβέλεια και η επιρροή αυτής της συμφωνίας και στα πλαίσια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα μας οδηγούσε να ξαναδούμε λίγο το ρόλο και του Ευρωπαίου Πευθύνου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εδώ σημαντικό είναι να επισημάνουμε ότι προβλέπονται μέσα στη συμφωνία μορφές συνεργασίας αυτόβουλες που αφορούν συγκεκριμένα κράτη-μέλη και είναι δραστηριότητες που συμπληρώνουν τις εθνικές εφόσον ισχύουν και η ισχύ στην η εδαφική ισχύ στον, της συμφωνίας είναι σαφής θα πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνίας, οπότε και από αυτήν την προοπτική είναι πολύ συγκεκριμένη και ακριβής και βεβαίω πολύτιμη η εντατικοποίηση των σχέσεων με την Ιαπωνία. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτά τα σχόλια να περιοριστώ προ στιγμή και να ακούσω και τι παρεμβάσει των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο. Σχόλια. Κύριε Μποζούτιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιακολίνο για την παρουσίαση και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο του. Την τελευταία φορά που ε, εξετάσαμε συμφωνία που είχε υπογραφεί 30, ε, ε, Νοεμβρίου, είχε υπογραφεί 30 Νοεμβρίου λίγο πριν τη θέση σε ισχύ τη ε, συνθήκη Λισαβόνα, το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία δεν πήγε καλά και ξέρουμε τι συνέβη. Α ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί το ίδιο και με τη συμφωνία αυτή με την Ιαπωνία, που, όπω είπε ο κύριο Γιακολίνο, είναι τεράστια σημασία χώρα και όπου, με την οποία ε, η συνεργασία πρέπει να ενθαρρύνεται και να στηρίζεται. Τώρα, επί τη βάση των πληροφοριών που μας έδωσε η Προεδρία και την ευχαριστώ, θα κάνω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών για τις τραπεζικές συναλλαγές και κινήσεις, σε ποιο βαθμό ε, εξετάζουμε μια συμφωνία δεύτερη τύπου SWIFT. Μπορεί να μας διαβεβαιώσουν ότι δεν μιλάμε για κάτι που θα μοιάζει με το SWIFT. Δεύτερον, για τις παρατηρήσεις σχετικά με τη θανατική ποινή. Αν κατάλαβα καλά, η διάταξη εδώ, όπως εξηγήθηκε από την Προεδρία, αναφέρεται σε μία υπόσχεση που έδωσαν οι Ιαπωνικές αρχές ότι θανατική ποινή δεν θα εφαρμοστεί σε πρόσωπα ε, που καλύπτονται από την ε, συμφωνία ή ε, επί των οποίων δίδονται πληροφορίες στα πλαίσια της συμφωνίας. Πρόκειται απλά για μια συμφωνία γιατί αυτό άκουσα από τη διερμηνία. Ανησυχώ λίγο όμως αν μόνο υποσχέσεις ελάβαμε και όχι νομική δέσμευση. Θα ήθελα παρακαλώ η Προεδρία να μου το διευκρινίσει αυτό. Άλλες παρεμβάσεις, κάποιος συνάδελφος άλλος που θέλει, ζητεί το λόγο. Δεν υπάρχουν. Επιστρέφομαι λοιπόν στην Προεδρία η οποία θα απαντήσει στις ε, παρατηρήσεις του κυρίου Μπουσουτήλ. Η Ισπανική Προεδρία. Ε, ε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας Πρόεδρε, αλλά και τον κύριο Μπουσουτήλ για τα σχόλιά του και τις παρατηρήσεις του. Θα ήθελα καταρχήν να επισημάνω ότι οι συμφωνίες Συνήθισε 30 Νοεμβρίου. Για τον το λόγο ότι οι διαπραγματεύσεις του άρχισαν πριν από μία διετία περίπου. Ξεκίνησαν πρώτα κάποιες άτυπες συνομιλίες, άρχισε τις διαπραγματεύσεις η Τσεχική Προεδρία, τη συνέχισε και τις διεκπαιρέωσε η Σουηδική. Αν περιμέναμε μετά τις 30 Νοεμβρίου, τότε η διαπραγματευτική εντολή θα εξέπνε. Οπότε θα έπρεπε να γίνει διαπραγμάτευση νέας εντολής. Κάτι που θα οδηγούσε σε καθυστέρηση. Εξηγήσαμε λοιπόν στην Ιαπωνία ότι για εσωτερικούς λόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη η διαπραγματευτική διαδικασία της διετίας δεν θα έπρεπε να καθυστερήσει άλλο, γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μία ανάγκη έναρξης εκ του μηδενός των διαπραγματεύσεων, αν είχαν ξεπεραστεί 30 Νοεμβρίου, κάτι που δεν θα μπορούσε να καταλάβει, να κατανοήσει η Ιαπωνία. Επαναλαμβάνω, μία καθυστέρηση της συμφωνίας θα οδηγούσε σε απέτηση για νέα διαπραγματευτική εντολή. Αποτέλεσμα να επηρεαστεί μια τρίτη χώρα, η Ιαπωνία, για λόγους που ήταν εσωτερικοί θεσμικοί λόγοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το SWIFT για τις τραπεζικές πληροφορίες, αυτό είναι μια απλή σύμπτωση. Δεν πρόκειται για γενική ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά για συγκεκριμένες αιτήσει χορήγησης πληροφοριών για τραπεζικούς λογαριασμούς που μπορεί ε, ένας εμπλεκόμενος σε μια διαδικασία να έχει. Πρόκειται για αιτήσει δικαστικής συνεργασίας που συνήθως γίνονται μεταξύ των χωρών μελών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το μεταξύ χωρών μελών και τρίτων χωρών. Σε ό,τι αφορά τη θανατική ποινή, Θα ήθελα να πω ότι ίσως δεν ήμουν αρκετά σαφής. Δεν ήταν α, ε, υπόσχεση αυτό που έδωσε η, η Ιαπωνία, αλλά δέσμευση, νομική υποχρέωση των Ιαπωνικών αρχών. Δεν είναι μία απλή υπόσχεση. Είναι μία νομική υποχρέωση που απορρέει από τη Συμφωνία. Νομική υποχρέωση που προκύπτει από το άρθρο 11 1 παράγραφο Β τη ε, συμφωνία Δικαστική Συνδρομή με την Ιαπωνία. Δεν ήταν απλή υπόσχεση, αλλά δέσμευση και νομική υποχρέωση που απορρέει από αυτό το άρθρο 11.1 Β. Σα ευχαριστώ. Κύριε Γιακολίνο, θέλετε να προσθέσετε ως ε, εισηγητής τελικά σχόλια. Ε, άκουσα με μεγάλη προσοχή και τις απαντήσεις της Ισπανικής Προεδρίας παρόλο που φαίνεται να ε, μην έλαβε υπόψη την παρατήρηση που έκανα και που θα τη διαβέσω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 18, αυτό που είπε και ο κύριος ε, Μπουσουτήλ για τις τραπεζικές συναλλαγές. Για να εξακριβωθεί και η αρχή της αναλογικότητας. Αν σε τέτοια περίπτωση περιλαμβάνεται και ο εγγυητής. Αυτή ήταν η μόνη παρατήρηση που έκανα εγώ. Και κατά του λοιπού το κείμενο είναι αρκετά σαφές. Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία που συνήθει με την Ιαπωνία και αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να την στηρίξουμε με τη λήψη συγκεκριμένη απόφαση. Ευχαριστώ κυρία Κολίνο. Uh, Εξαντλήσαμε και αυτό το θέμα της σημερινής διάταξης που περιλάμβανε απλώς παρουσίαση της ε, έκθεσης και είμαστε έτοιμοι για την συνέχεια της διαδικασίας. Αφού περάσουμε στα διάφορα και διεκπαιρεώσουμε και το σημείο 18, μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας. Αν δεν υπάρχουν διάφορα λοιπόν, η ημερομηνία της προσεχούς συνεδρίασης έχει καθοριστεί η 7η Απριλίου από τις 9 με 12.30 και 3 με 6.30 και 8 Απριλίου 9 με 12.30. The afternoon of the 7 Το απόγευμα της 7ης Απριλίου η συνεδρίαση δεν θα αρχίσει στις 3 αλλά στις 4.30 γιατί θα έχουμε μείνει ολομέλεια Γι' αυτό και η συνεδρίαση απογευματινή της 7ης Απριλίου θα ξεκινήσει 4.30 μέχρι τις 8.